La Άρχεται η σύνοδος. Καλημέρα σας. Come Όπως γνωρίζετε, πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, σήμερα το πρωί, είναι ο εορτασμό τη 10η επαιτίου τη συνθήκη τη Λισαβόνα και του νομικά δεσμευτικού χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να θυμίσω στους βουλευτές ότι για αυτήν τη συζήτηση δεν θα έχουμε το, τη διαδικασία ε, προσέλκυσης προσοχής του Πρόεδρου. Ούτε ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ για να ορτάσουμε μαζί την δέκατη επέτειο από την θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας και της ε, νομικά, του νομικά δεσμευτικού χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πέρσι, την 1η Δεκεμβρίου, σε μια τελετή στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ε, με παρουσία των κυρίων Μισελ, Λαγκάρτ και Φοντερ Λάιεν θελήσαμε να θυμηθούμε αυτήν την συμβολική επέτειο και να ξεκινήσει και ένας ε, νέος θεσμικός κύκλος για τη νέα θητεία ε, σήμερα. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε ότι περνώντας για το Στρασβούργο περνάμε και από τη Γερμανία και διασχίζουμε ένα σύνορο χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Ένα σύνορο που το 1860 το 1870 βάφτηκε με αίμα. Ε, γενναίες ε, Ευρωπαίων έχουν ζήσει αυτή τη φάση. Τώρα μπορούμε να περνάμε ειρηνικά και είναι μια μεγάλη κατάκτηση αυτή. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, ιδίω σήμερα που εορτάζουμε τα 75 ε, χρόνια. 75 χρόνια από τη μάχη των Αρδενών που ε, οδήγησε στο θάνατο νέων Ευρωπαίων, ε, χιλιάδων νέων Ευρωπαίων και σημάδεψε εκείνες τις γενιές. Πρέπει να θεμόμαστε ότι το ευρωπαϊκό επίτευγμα είναι το μόνο που μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ένα χώρο ειρήνης ε, ε, ένα χώρο δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη. Και αυτό καλούμαστε να προσπιζόμαστε καθημερινά. Εργαζόμενοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να την κάνουμε ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική. Η θέση σε ισχύ ε, πριν από 10 χρόνια τη συνθήκη τη Λισαβόνα ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου για, τους, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και του πολίτε για τι χώρε μα και πραγματικά και για το Κοινοβούλιο για την ε, ευρωπαϊκή δημοκρατία, γιατί ενισχύεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας της Ένωσής μας, η αποτελεσματικότητά της, η διαφάνειά της και αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο για τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν πλέον να εκφράσουν τη φωνή τους χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ και δέκα χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο συνεγκρίνουν τον ε, τήσιο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αποφασιστικότερο ρόλο στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όμω να μην ξεχνάμε ότι πίσω από του αριθμού, τι δημοσιονομικέ γραμμέ και το δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν πάντοτε πρόσωπα, άνθρωποι. Και εκείνους ε, πρέπει να σκεφτόμαστε όταν αναζητούμε απαντήσει. Χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα μπορούμε να σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ε, ισότητα, την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και το κράτο δικαίου. Όλα αυτά έγιναν πυλώνε επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε ε, νομικώ δεσμευτικούς κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη και όλα τα θεσμικά όργανα. Παρόλα αυτά, οι διακρίσεις συνεχίζονται και πλήττουν τις χώρες μας. Οι ειδήσει μας θυμίζουν διαρκώς ότι η βία κατά των γυναικών, ο ρατσισμό, οι διάφορες μορφές ε, έλλειψης ανεκτικότητας, αυτή τη στιγμή πραγματικά οδηγούν σε άθλιες συνθήκε πολλού Ευρωπαίους Και με την Παγκόσμια ημέρα της ε, αλληλεγγύης ε, πριν από λίγες μέρες ε, πρέπει να θυμίσω ότι θέλουμε μια Ευρώπη ελευθερότερη και πιο ίση. Θέλουμε να σκεφτόμαστε το κοινό μας μέλλον όλοι μαζί και πρέπει να βαδίσουμε χέρι-χέρι. Χάρη στη μεγάλη συμμετοχή στι πρόσφατε εκλογέ, οι πολίτε μα μας μετέφεραν ένα σαφέ μήνυμα. Θέλουν να συνεισφέρουν περισσότερο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είμαι πεπισμένος ότι η Σύνοδος για το μέλλον της Ευρώπης που σκοπεύουμε, η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης που σκοπεύουμε να, να οργανώσουμε τις επόμενους μήνες θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γι' αυτό. Ε, πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες με αφορμή αυτή τη διάσκεψη, τις απαιτήσει τους ε, και τις ελπίδες τους και να ε, προβλέψουμε μια καλύτερη, ευρυθμότερη λειτουργία του δημοκρατικού μας συστήματος. Είναι καθήκον μας να μεταφράσουμε στην πράξη τις απαιτήσει και τις επιθυμίες των πολιτών και να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας όλη αυτή η, ε, όλο αυτό το εγχείρημα. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτελεσματικότερο τρόπο να αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Όλα αυτά βέβαια, όλες αυτές οι προθέσεις και οι προτάσεις θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομοθετικές κοινοβουλευτικέ πράξεις και ενέργειες και πολιτικές δράσεις. Νομίζω ότι η γενιά μας μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον πρόεδρο Μάνφρεντ Βέμπερ. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ας το καταλάβουμε. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας Ήρθε η Ευρώπη να επανορθώσει όσα πέτυχε όταν επιχείρησε να ε, ε, βρει ένα σύνταγμα. Μαθαίνουμε από τα σφάλματά μας και χάρη στις κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε μια ένωση έκανε την κοινότητα ένωση. Έδωσε ένα πολιτικό πρόσωπο στην Ευρώπη για να έχει μία φωνή στην εξωτερική πολιτική. Ε, Καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι με παγκόσμιους ηγέτες. Ε, ας πούμε και στο θέμα της συμφωνίας με το Ιράν. Ενίσχυσε το ρόλο των πολιτών. Η συναπόφαση έγινε ε, ο κομβικός τρόπος ε, νομοθέτησης στην Ευρώπη. Σήμερα το κοινοβούλιο μας έχει ισχύ και επίσης Έχουμε και νέε αρμοδιότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταπολέμηση του εγκλήματο, η ανταλλαγή δεδομένων, η πολιτική ασύλου. Όλα αυτά έγιναν ευρωπαϊκά ζητήματα και έφεραν περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη ενεργητική και παθητική. Επίση, ε, έδωσε η συνθήκη τη Λισαβόνα δεσμευτικό χαρακτήρα στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατοχύρωσε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Αυτό μα λέει ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι σημαίνει να ε, είσαι, να Ευρωπαίο. Ε, κράτους δικαίου, δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η Ευρώπη δεν πήγαινε ποτέ ευθεία, δεν ήταν ποτέ ευθεία η πορεία της. Με μικρά βήματα προχωρούσε. Η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ένα άλμα προς ένα σύγχρονο τρόπο ε, συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η Εύλιν Μπέρκ είχε πει ότι ένα κράτος που δεν μπορεί να αλλάξει είναι ένα κράτος που δεν μπορεί να συνδιαλέγεται και να συνομιλεί. Ε, τώρα έχει ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, ας πάμε στα επόμενα. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι καταπληκτική ευκαιρία. Όπως είχε πει ο Στεν, όταν κήρυξε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, τότε της Συντακτικής Συνέλευσης, είπε ας ονειρευτούμε την Ευρώπη. Εγώ θα πω ας ξανά ονειρευτούμε την Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσουμε θεμελιώδη ερωτήματα. Ποια είναι τα βασικά πεδία όπου θα πρέπει να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά να δράει η Ευρώπη όπου έχει προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή για τους πολίτες. Ακόμα ε, παραμένουν κάποια ε, πεδίο που χρειάζεται η Ευρώπη τα σωστά εργαλεία για να δρά. Ένα δεύτερο θέμα για το μέλλον. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι ακόμα ανοιχτό. Διότι οι πολίτες θα εμπιστευθούν την Ευρώπη μόνο ε, όταν λογοδοτούν όσοι λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Και το τρίτο είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρώπης και να αντέξουμε στη σύγκρουση Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών γιατί κινδυνεύει η Ευρώπη να χαθεί αν δεν έχει μια φωνή. Ας γράψουμε τώρα μαζί την ευρωπαϊκή ιστορία αφού γραζόμενοι τους πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως εκλεγμένο σώμα. Εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ομάδας μας έχουμε μια σαφή ιδέα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι ε, ο ε, ελάχιστος κοινό παρονομαστής, ένα άθροισμα ιδεών, μια γενική και όριστη άσκηση Θέλουμε κάτι ουσιαστικό και όχι κάτι τεχνικό για την Ευρώπη. Μια ουσιαστική και γνήσια συζήτηση. Τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος για να ε, δημιουργήσουμε δίπλα στην εθνική ταυτότητα του καθενός και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ας είναι αυτή η επέτειος λοιπόν η δεκαετής η αρχή ενός νέου ευρωπαϊκού ονείρου. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ομάδα του είναι έτοιμο να κάνει τη διαφορά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος Γκαρθία Πέρες. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέκα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας έχουμε μια καλή ευκαιρία για απολογισμό. Μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή ήταν ε, μια επιτυχία της τότε Προεδρίας της Πορτογαλικής με σοσιαλιστική κυβέρνηση σε μια στιγμή πάρα πολύ λεπτή. Θυμάστε τι ε, τραύμα ήταν η απόρριψη του του Ευρωπαϊκού Συντάγματος το 2005 από δύο κράτη-μέλη και η αβεβαιότητα που δημιούργησε αυτό. Ωστόσο, ακολούθησε ε, ε, συνέχεια. Δεν ήταν μάταιη η εργασία της ε, συντακτικής συνέλευσης το 2002 το 2003. Οι ευρωπαϊκές κοινότητες είχαν επικεντρωθεί πάρα πολύ στα θέματα της αγοράς και τα οικονομικά και είχαν ξεχάσει τις φιλοδοξίες. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ε, που να είναι ικανή να λύνει τα προβλήματα των πολιτών. Ήταν σωστό να ασχοληθούμε με θέματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η Ευρώπη των πολιτών και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ωστόσο, τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις κάτω χώρες έδειξαν ότι κάποιοι από τους πολίτες τουλάχιστον δεν θεώρησε ότι είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Ευτυχώς κάποια σημαντικά στοιχεία μπήκαν στη συνθήκη της Λισαβόνας και έγιναν σημαντικά βήματα πρόοδου. Από τη μια Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί να προσχωρεί σε συνθήκες και συμβάσεις διεθνούς χαρακτήρα και επίσης έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας και έχει βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι νομικά δεσμευτικός και επίσης έχουν ενισχυθεί τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αρκεί αυτό, άρα προφανώς όχι. Προφανώ οι πολίτε, άνδρε και γυναίκε, περιμένουν περισσότερα από εμά. Εξού και η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη είναι μια ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να χαθεί. Για να δοθεί νέα πνοή, νέα όθηση ε, στη διαδικασία ολοκλήρωση, να είναι πιο δημοκρατική και πιο κοντά στον πολίτη. Α μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντο. Θα πρέπει να υπολογίζουμε και να ποντάρουμε στου πολίτε από την αρχή, να αισθάνονται ότι συμμετέχουν. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσει ερήμην των πολιτών. Αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα με τη συνθήκη. Υπάρχει περιθώριο. Για παράδειγμα, να ε, κατοχυρώσουμε το σύστημα του επικεφαλής, του κορυφαίου υποψηφίου ή τα υπερεθνικά ε, ψηφοδέλτια στις ευρωεκλογέ. Να σταματήσει η παράλυση της ομοφωνίας ε, όπως, σε θέματα τόσο κομβικά όπως είναι η φορολογία, η εξωτερική πολιτική, για να έχουμε μια δίκαιη φορολογία και να ξεπερνάμε το μπλοκάρισμα στη διεύρυνση, ας πούμε, όπως τώρα με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Δεν έχουμε ούτε στιγμή να χάσουμε εδώ. Το γνωρίζουν αυτά τα μέλη του Συμβουλίου και γι' αυτό την περασμένη εβδομάδα κατάφεραν να ξεπεράσουν άτυπα την ομοφωνία για να εγγυηθούν την ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα πριν το 2050. Ας ελπίσουμε να μην μείνει μόνο σε αυτά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μειώσει, να αποφασίσει να μειώσει του τομεί όπου χρειάζεται ομοφωνία. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που έχουμε. Α αρχίσουμε τώρα ένα ε, νέο πολιτικό κύκλο. Τώρα έχει έρθει η ώρα να επιδείξουμε θάρρο. Έχει αλλάξει η Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την κλιματική έκτακτη ανάγκη, για την έμφυλη βία, για του πρόσφυγες που κρούν τι θύρε τη Ευρώπη που ψάχνουν να βρουν μια μοίρα και ένα μέλλον, την παιδική φτώχεια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Α ασχοληθούμε σοβαρά με αυτή την ευκαιρία και με του πολίτε και την κοινωνία των πολιτών για να γίνει η Ευρώπη μα και καλύτερη και ισχυρότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Πασκάλ Τυρό για την Renew Europe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε και εσεί ε, στην ομιλία σα όταν αναλάβατε και ξέρετε ότι αναλαμβάνετε καθήκοντα πολύ σοβαρά. Είναι μια εποχή ωραία. Στην Γαλλία τα παιδιά πάνε από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Περνάμε σε μια νέα εποχή, σε, μια, ε, σε νέους καιρούς. Ε, και τα παιδιά αναλόγως πηγαίνουν από την άνεση του δημοτικού σχολείου σε μια κατάσταση πιο ε, απαιτητική. Ο κόσμο έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα χρόνια. Το ξέρετε κι εσεί και το ξέρουμε κι εμεί. Οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα δεν είναι οι ίδιε με αυτέ που είχαμε πριν από δέκα χρόνια. Τα κλιματικά προβλήματα, τα κοινωνικά, το θέμα τη μετανάστευση και τη μετακίνηση των πληθυσμών, τα δημογραφικά. Ο κίνδυνο που βαραίνει τι δημοκρατίε μα, που πολλέ φορέ είναι στο εσωτερικό τη Ένωση, το κράτο δικαίου. Όλα αυτά είναι θέματα. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα να εξελιχθούν. Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο πρέπει και εμεί να αλλάξουμε του δικού μα κανόνε και πρέπει αυτό να γίνει στη λογική της δημοκρατίας και του σεβασμού του κράτου δικαίου. Το λέω και στρέφομαι προς το Συμβούλιο. Η διακυβερνητική μέθοδος πρέπει να αλλάξει πρέπει επιτέλους να επαφίεστε περισσότερο στην εκπροσώπηση και την αντιπροσώπευση των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή το Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προόδου και είναι καθοριστικό. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και το Συμβούλιο το ίδιο πρέπει να γίνει διαφανέστερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε θα μπορεί να βασίζεται σε δύο συνομοθέτε. Και όπω ε, το είπαμε και η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, που εσεί ε, αναφέρατε στην ομιλία σα, κυρία Πρόεδρε, είναι κάτι το ουσιαστικό. Το θέλουμε. Σε δέκα χρόνια θέλουμε οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών να ε, ε, συνεχίσουν όπως έγινε να παίρνουν μέρος στις δημόσιες συζητήσεις και θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει χωρίς του πολίτε, χωρί την κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η διάσκεψη για την Ευρώπη δεν θα πρέπει να αρκεστεί στο να ακούει απλώ του πολίτε. Πρέπει να έχουν συμμετοχή, να χτίσουν μαζί μα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και να μην είναι απλώς το άθροισμα 27 εθνικοτήτων, υπηκοτήτων των 27 κρατών μελών. Υπάρχει κάτι που τα, που τα υπερβαίνει όλα αυτά το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ε, ξέρω, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι στο πλευρό σα, ώστε οι πολίτε, η κοινωνία των πολιτών, να πάρουν μέρο στι δημόσιε διαπραγματεύσει και συζητήσει. Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να περάσει. Είναι ε, μοναδική και επιτέλου η Ευρώπη μπορεί να έρθει κοντά στου πολίτε τη. Και θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Πριν από 70 χρόνια, Είχαμε ένα άλλο ε, σημαντικό γεγονό. Ο κύριο Τσέρτσιλ στην πλατεία Κλεμπέρ βγήκε σε ένα μπαλκόνι και ε, εκφώνησε μια ομιλία. Και θέλω να σα αναφέρω κάτι από αυτά που σε εκείνη την ομιλία. Οι κίνδυνοι που μα απειλούν είναι μεγάλοι. Αλλά μεγάλη είναι και η δύναμή μα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην επιτύχουμε και να μην επιτελέσουμε το στόχο μας, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα οικοδόμημα, μια έννοια Ευρώπη. Αυτό υπόθηκε πριν από 70 χρόνια και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε Λάμπερτ, Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο μέχρι, μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, με την πρόοδο στην οικοδόμηση αυτής της ε, ε, δημοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αυτό που είναι. Ε, χωρίς τη Λισαμβόνα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λόγο στις διεθνείς συνθήκες και να, είμαστε, να συνυπογράφουμε ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να έχουμε βασικούς ε, υπεύθυνους όπως αυτούς που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Λισαμβόνα λοιπόν ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων έγινε υποχρεωτικός νομικά έτσι ώστε η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, ε, η ιδιότητα του πολίτη, η δικαιοσύνη ε, για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να διασφαλιστεί. Πολλοί από τους ε, συμπολίτες μας ε, βέβαια, ειδικά στην Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία, ε, είδαν στην αρχή την συνθήκη της Λισαβόνας ως άρνηση της δικής τους κυριαρχίας. Όμως, μια νέα συνθήκη φαινόταν κάτι ως, ένα νεοφιλελεύθερο εγχείρημα που θα εμπόδιζε τις δημόσιες επενδύσεις. Όμως, ε, φαινόταν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, κεφαλαίων επίσης θα ήταν πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ε, φαίνεται ότι τελικά τα κοινωνικά δικαιώματα που συχνά τα κράτη δηλώνουν στις προθέσεις τους τώρα διασφαλίζονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να αποδοκιμάσει τις συνθήκες ε, που θεωρούσε ότι δεν ήταν ε, σωστές, όπως ε, η συνθήκη με το Μερκοσούρ, που θα μπορούσε να επιδεινώσει το περιβαλλοντικό σύστημα. Επίσης, στην κοινή αγροτική πολιτική, στην απόφαση, εμείς μπορέσαμε να καταθέσουμε νέες προτάσεις στην Κομισιόν που τελικά οδήγησαν στο Green Deal. Κυρία Φοντερ Λάινεν, έτσι έχουμε μία πόρτα η οποία δεν θα μπορέσει να μας ε, επιτρέψει να ε, παρακάμψουμε ε, σε, νομικά, σε φορολογικά θέματα το Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε θαραλέοι, γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών μας είναι που θα μας ανταμείψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τζάνι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα θα καλούμαστε να ρωτάσουμε τη δεκαετή επέτειο μια συμφωνία που θα έπρεπε να έχει οδηγήσει και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μέλλον ανάπτυξη και ευημερία. Ωστόσο, τα γεγονότα δυστυχώς ε, αποδεικνύουν ότι αυτή η συμφωνία πέτυχε. Σήμερα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο αδύναμα. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πιο ευπαθείς και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια βαθιά θεσμική και πολιτική κρίση. Αυτό πραγματικά αποδεικνύει περίτρανα ότι απέτυχε παταγωδός μία προσέγγιση κεντρικού, κεντρική οργάνωση ε, που ήθελε να φέρει η συνθήκη τη Λισαβόνα, να αποφασίζουν τα κράτη χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών ε, εθνών, ευρωπαϊκών κρατών. Αυτά εδώ τα αντιλαμβάνεστε ω ε, κίνδυνο, όμω θα πρέπει να είναι αξίε που προστατεύονται. Σήμερα βλέπω να υπάρχουν ομοιότητες σε σχέση με την προσέγγιση του παρελθόντος και ετοιμάζεστε να διαπράξετε, να διαπράξετε τα ίδια σφάλματα που το Συμβούλιο με τον προκάτοχο του κυρίου Μισελ ε, διέπραξε με το σφάλμα του δημοψηφίσματος του Brexit. Τότε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έδειχναν μια αποστροφή σε σχέση με το αίσθημα που εξέφραζαν κάποιοι ευρωπαϊκοί λαοί. Το ίδιο λάθος ε, έγινε με το Brexit και το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Ε, όμως πραγματικά μπορέσαμε με τρόπους ε, ε, υπόγειου και διπλωματικού να αποφύγουμε το αποτέλεσμα του Ιρλανδικού τότε δημοψηφίσματο. Όχι όμω και του Βρετανικού. Ε, αυτό που ήταν η κυρίαρχη επιλογή και η απόφαση του Βρετανικού λαού το 2016. Η συμβουλή μου προ το Συμβούλιο λοιπόν να μην διαπράξετε τέτοιο σφάλμα. Ε, τώρα θα βρεθούμε από το Γενάρη να πρέπει να διαπραγματευτούμε μια σημαντική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και η προσέγγιση που θα ακολουθήσει το Συμβούλιο και το δικό μα σώμα δεν θα πρέπει να είναι προσέγγιση τιμωρητική κριτική προ του Βρετανού πολίτε για την επιλογή του. Θα πρέπει ε, να μην προσπαθούμε να ανατρέψουμε μια δημοκρατική απόφαση ενό λαού του Βρετανικού, αλλά να εργαστούμε για μια συμφωνία που θα προστατεύσει τι επιχειρήσει μα, τι εταιρείε μα, αλλά κατ' επέκταση και του πολίτε μα. Και θα ε, μα επιτρέψει και μετά το 2020 να έχουμε μια σχέση ε, εποφελού συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι σε θέση να αφουγκραστούν περισσότερο τις ανάγκες των πολιτών και να λάβουν υπόψη τις ε, αποφάσεις τους καθώς και τις κυρίαρχες αποφάσεις των 100 μελών, τότε ούτε σε άλλα 10 χρόνια δεν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε την 20η επέτειο από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστούμε ο κύριος Τζαμπάσκι. госпожо господин Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 10 χρόνια από τη συνθήκη της Λισαβόνας, από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι μια συνθήκη η οποία θα έπρεπε να δημιουργήσει μια συνταγματική Ευρώπη, όμως ήταν και ένας από τους λόγους που η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ε, θεσπίστηκε στην Ευρώπη εμείς ε, είχαμε αξίες που υπερασπιζόμασταν που δεν συνείδαμε ε, τα υπόλοιπα. Θέλαμε περισσότερη διαφάνεια, θέλαμε περισσότερη δημοκρατία, να μην υπάρχει τόσος κεντρικός έλεγχος, να υπάρχουν πιο πολλές κοινέ αποφάσεις. Ε, οι άνθρωποι γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν να μην ε, εμπιστεύονται τη δουλειά των θεσμών. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι και ένας από τους λόγους για το Brexit. Υπάρχουν εδώ σε αυτή την αίθουσα σήμερα άνθρωποι ακόμα που συνεχίζουν να επιτίθενται σε κράτη-μέλη και σε κυβερνήσεις ε, που είναι νόμιμα εκλεγμένες. Θέλουν να τιμωρήσουν τα κράτη-μέλη για τις κυρίαρχες αποφάσεις τους π.χ. σε θέματα μετανάστευσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν όμως αυτός ο πραγματικός σκοπός. Εγώ θέλω να πιστεύω πως δεν ισχύει αυτό. Δεν πιστεύω στο σούπερ κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Δεν ε, θέλω να πιστεύω ε, ότι αυτό θα αντικαταστήσει τη δική μου χώρα. Η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ένα λάθος. Ήταν μια προσπάθεια συμβιβασμού, όμως οδήγησε και σε, στη λάθος μορφή ε, ομοσπονδιοποίησης. Η Ευρώπη είναι, απαρτίζεται από κράτη-μέλη που πρέπει να δείχνουν αμοιβαίο ε, σεβασμό και να προχωρούν μαζί. Καλές διακοπές σε όλους για να καταλήξω. Κυρία Ομπρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περίεργη αίσθηση για μας η ε, εορτασμή αυτή ε, της επαιτίου τη συνθήκη Λισαβόνα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί μετά από τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων σε Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία. Έδειξε πόσο αντιδημοκρατικά είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο επάταξαν την Ελλάδα. Τώρα έχουμε την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες η επισύναψη του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στη συνθήκη δεν ε, βοηθάει την κατάσταση, γιατί δυστυχώς αυτό παραμένει φιλοσικής ε, σε μια αγορά άκαρδη δυστυχώς δεν είναι λόγος Θεού η συνθήκη. Μπορεί κανείς να την αφισβητήσει. Η νέα πράσινη συμφωνία, η κοινωνική και η οικολογική, δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ με την ισχύ που θα έπρεπε με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο. Η μετάβαση ε, οικολογική περιορίζεται και ε, φρενάρεται από το χρυσό κανόνα για τα δημοσιονομικά. Τώρα καταστρέφουν και τις συντάξεις μας και αυτό το προωθεί και το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιστορική απόφαση αυτή την εβδομάδα. Ε, βλέπουμε ένα γενικό dumping, το οποίο ενθαρρύνεται από το δόγμα των ελεύθερων συναλλαγών και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη όσο παραμένουν φορολογική παράδειση και έχουν και βέτο το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. Ε, αυτά όλα λοιπόν είναι προφάσεις αναμαρτίες. Χάνουμε χρόνο. Ενώ θέλουμε ε, μια επανάσταση να κινητοποιήσουμε ε, μεταπολεμική. Θα πρέπει το παρελθόν παρελθόν να ε, αναθεωρηθεί εκ βάθρων με τη διάσκεψη για την Ευρώπη. Δημοκρατική με υποχρεωτική συμμετοχή των λαών. Δικαίωμα πρωτοβουλία ε, του Κοινοβουλίου. Μηδενική ανοχή στα λόμπι. Διαφάνεια στο Συμβούλιο Ένα πράσινο κανόνα που να προστατεύει του φυσικού όρου με καθολική πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, με ε, προστασία κατοχυρωμένη των κοινοφελών υπηρεσιών και όχι καταστολή ε, φορολογική και κοινωνική. Θα πρέπει να είναι ένα σύμφωνο προόδου, αρμονικό και βιώσιμο και όχι σύμφωνο ανάπτυξη και σταθερότητα. Μόνο έτσι θα έρθει η νέα πράσινη συμφωνία και μόνο έτσι θα συμφιλειωθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί με την ίδια την ιδέα τη Ευρωπαϊκή συνεργασία. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τι έκτακτε καταστάσει του παρόντο. Αυτά θα πρέπει να είναι τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε στη δεκάτη επέτειο τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπο... Κύριος Μπόλοκ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αν δεν υπήρχε η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε το Brexit σήμερα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που εσείς αποφασίσατε να επεκτείνετε τις δικές σας εξουσίες να φτιάξετε ένα σούπερ κράτος και αγνοήσατε τη δημοκρατία των εθνικών κρατών όπως και τους ψηφοφόρους. Το εργατικό κόμμα τότε δεν μας έδωσε δημοψήφισμα και τώρα μάλλον το μετανιώνουν. Και η Ιρλανδία φυσικά έκανε ε, δημοψήφισμα, δεν έβγαλε καλό αποτέλεσμα και έπρεπε να ξαναψηφίσει. Αυτό που είπε η Μάργαρετ Θάτσερ ε, στο παρελθόν ήταν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ένας θεσμός ο οποίο ε, τελικά έχει φτιαχτεί για να μετατρέπεται συνεχώ σύμφωνα με κάποιες αφηρημένε πνευματικές ε, ε, ιδέες. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, είπε η Θάτσερ, όμως αυτό έγινε. Στην συνθήκη της Λισαβόνα έχουμε το άρθρο 30 και υπάρχουν και μέσα για να φύγει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν παγίδα. Η Βρετανία όμω κατάφερε να ψηφίσει και να ελευθερωθεί από αυτό χάρη στην πίεση του και του του Brexit που οδήγησε σε μία μεταρρύθμιση στο πάρτι στο κόμμα των Τόρις και, και τον Μπόρις Τζόνσον θα μπορέσουμε τελικά ε, να φύγουμε έτσι. Μπορείτε κι εσείς να γιορτάσετε τη δική σας συνθήκη και εμείς να γιορτάσουμε τη δική μας κυριαρχία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία ως ελεύθερη χώρα για άλλη μια φορά. Ε, και ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην πρόεδρο Φόντερ Λάιον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όταν ε, κοιτάμε την αρχή του αιώνα, ε, Κάτι έλειπε ε, στο ευρωπαϊκό ε, εγχείρημα. Είχε πέσει ήδη το σιδηρούν παραπέτασμα. Οι ευρωπαϊκές κοινότητες ε, ήταν ήδη μία καλά εγκατεστημένη πραγματικότητα, όμως κάτι έλειπε. Όπως είπε ο προκάτοχός μου Ζακ Ντελόρ, η Ευρώπη χρειαζόταν μια ψυχή. Είχε πει ήρθε η στιγμή να δώσουμε μια ψυχή στην Ευρώπη. Αυτό έκανε η Λισαβόνα. Αν ρωτήσετε τους δικηγόρους θα σας εξηγήσουν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην Ευρώπη μια ενιαία νομική προσωπικότητα. Ναι, φυσικά, αυτό έγινε. Όμως έγινε και κάτι παραπάνω. Έδωσε στην Ευρώπη μια ψυχή ή μάλλον την βοήθησε να ανακαλύψει και πάλι την πραγματική της ψυχή. Αυτή η ψυχή μας έκανε να πατάξουμε την τυραννία, να την νικήσουμε. Έφερε, ε, ε, ε μας οδήγησε στο να καταρρεύσει το σιδηρούν παντραπέτασμα και να ξαναενωθεί η Ήπειρός μας. Η, η συνθήκη της Λισαβόνας είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιώματα και ελευθερίες για όλους. Έδωσε επίσης ένα κεντρικό ρόλο στους πολίτες της Ευρώπης. Έδωσε εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ο οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Επίσης έφερε τα Εθνικά Κοινοβούλια στο προσκήνιο και έδωσε στους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να ζητήσουν από την Κομισιόν να προτείνει νομοθεσίες. Ήταν μια ανάσα καθαρού αέρα στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ναι, δημιουργήθηκε γύρω από την οικονομία. Όμως η Ευρώπη πάντοτε είχε, έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από ότι ο άνθρακας και ο χάλιβας, από ότι μια ενιαία αγορά. Πάντοτε ε, προοριζόταν να είναι μια ένωση. Με την Λισαβόνα αυτό το σκοπό ξανανακαλύψαμε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε δύσκολους ανέμους που φύσηξαν ε, στην Ένωσή μας. Όμως, εμείς είμαστε σαν το καλάμι που λυγίζει αλλά δεν σπάει. Οι νέες προκλήσεις δεν, δεν την παραλύουν, την βοηθούν να προχωρήσει. Γιατί ε, χρησιμοποιεί ε, τις αρχές της και τις αξίες των συνθήκων της ε, για να θεμελιώσει τις ε, δυνάμεις της είναι ο λαός της Ευρώπης που τη στηρίζει. Η ένωσή μας δεν είναι ένα τετελεσμένο γεγονός, είναι μία αέναη δημιουργία. Και η οικοδόμηση είναι μία επιλογή που ανανεώνουμε κάθε μέρα. Είναι αυτό η ομορφιά της και η μοναδικότητά της. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι έχουμε, δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Από το 2016 όταν ήμουνα στη Γερμανία υπουργό ε, Άμυνας ε, είχα συνεισφέρει στην ανακάλυψη της ε, μόνιμης ε, διαρθρωμένης συνεργασίας στο θέμα της άμυνας. Ήταν ήδη στη συνθήκη, αλλά το δυναμικό της δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί. Η συνθήκη έχει πολλά ακόμα να μας προσφέρει. Για να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική, πιο δυνατή και πιο κυρίαρχη. Σε εμά τώρα πέφτει το βάρος ε, να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό της Λισαβόνας ε, και γι' αυτό είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα για να γιορτάσουμε τη δεκαετία επέτειο. Όσο το κάνουμε αυτό, κοιτάμε προς το μέλλον, προς τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα είναι αυτά τα χρόνια αυτό που εμείς θέλουμε να είναι. Θα είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες μας να κάνουμε. Την εποχή της Λισαβόνας ακόμα αναρωτιόμασταν αν η Ευρώπη μπορεί να έχει έναν ύμνο ή μια σημαία. Τα τελευταία δέκα χρόνια εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν κατέβει στους δρόμους κραδένοντας την μπλε σημαία με τα 12 αστέρια, τη δική μας ευρωπαϊκή σημαία. Υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι οι οποίοι με ενθουσιασμό ανακάλυψαν τις νότες του ύμνου στη χαρά τον εξαίρετο ύμνο της Ένωσής μας. Η Ευρώπη είναι οι πολίτες της. Γι' αυτό και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει και αυτή να είναι πάνω απ' όλα η δική τους διάσκεψη. Πρέπει να ακούσουμε αυτό που έχουν να μας πούν. Πρέπει να απαντήσουμε στις ανησυχίες τους, στις ελπίδες τους, γιατί αυτό αυτό είναι ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορούμε να αποτίσουμε στην συνθήκη της Λισαβόνας. Μία συνθήκη που έδωσε μια ψυχή στην Ευρώπη που δημιούργησε μία Ευρώπη των πολιτών, ε, μία Ευρώπη που έθεσε τους πολίτες στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρίσματος. Αυτή η Ευρώπη είναι το, η δική τους επιλογή, το δικό τους μέλλον. Είναι μια Ευρώπη που είναι δική μας επιλογή και που θέλουμε κάθε μέρα με πράξεις να την ανανεώνουμε. Ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Και τώρα εσείς Πρόεδρε Μισελ. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σα για να γιορτάσω τη δέκατη επέτειο από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο εορτασμό αυτό ε, απλώνει μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντο και του μέλλοντο τη Ευρώπη. Και πιο καλύτερο μέρο για να θυμηθούμε αυτό το ιστορικό γεγονό παρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα λαμπρό σύμβολο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Κυρίε και κύριοι, τα θεσμικά όργανα έχουν σημασία, διότι η νομιμοποίηση και η συνέχεια που χρειάζεται στο έργο του Ευρωπαϊκού εγχειρήματο, αυτό ακριβώς ε, είναι ακριβώς αυτό που προσφέρουν. Και Ακριβώς αυτό φαίνεται με τον εορτασμό το σημερινό, το τι εκπροσωπούμε. Α κοιτάξουμε λιγάκι το παρελθόν. Η συνθήκη της Ρώμης επιβεβαίωσε μια, με μια συνθήκη την ε, ε, υπόσχεση της Ευρώπης που ενώνει τα πεπρωμένα των ευρωπαϊκών λαών για πάντα. Η συνθήκη του Μάστριχτ θυμίζει την ιστορική σημασία του τέλους του κατακαιρματισμού της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ε, βοήθησε στην επούλωση των πληγών μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας έκανε τον νομικά δεσμευτικό χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ακριβώς αυτό, δεσμευτικό επέτρεψε να βασιστούμε σε ένα σύνολο κοινών αξιών. Δημιούργησε το σημερινό ευρωπαϊκό τοπίο, το οποίο βασίζεται σε αξίες και δημοκρατικούς θεσμούς, ε, ώστε να είμαστε σεβαστοί στο διεθνές προσκήνιο και ε, έχουμε, να αναλαμβάνουμε και να φέρνουμε σε πέρα στη δέσμευση να βελτιώνουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Πραγματικά είμαστε όλοι ταγμένοι στο σκοπό των θεμελιωδών ε, ε, δικαιωμάτων τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι ένα φωτεινό φάρο για να οδηγούμαστε προ την επίτευξη αυτών και την τήρηση αυτών των σοβαρών αξιών. Η συνθήκη τη Λισαβόνα ενισχύει την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου να νομοθετεί για την Ένωσή μα. Η συνθήκη τη Λισαβόνα επίση δίνει στην Ευρώπη μια ισχυρότερη φωνή στα διεθνή πράγματα και συγχρονίζει τι τοποθετήσει των ευρωπαϊκών κρατών και τι πολιτικέ του. Σήμερα μπορούμε να είμαστε πιο ενωμένοι ενώπιον του υπόλοιπου κόσμου. Και να, για να θυμίσω τα λόγια του Υπουργού Καρπίλτ, θέλω η Ευρώπη να είναι ε, ένας ε, παίκτη και όχι ένα άθυρμα, ένα παιχνίδι στα χέρια άλλων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ανυπομονούμε. Έχουμε πολλές προκλήσεις για το μέλλον. Το κλίμα, την ψηφιακή ατζέντα, την ειρήνη, την ασφάλεια, την άμυνα, την δυνατότητα να μιλάμε με μια ισχυρή ενωμένη φωνή στο διεθνές προσκήνιο περισσότερο από ποτέ συμμερίζομαι την ε, βεβαιότητα ότι έχουμε δίκιο να έχουμε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ε, ξεκινά μια νέα θεσμική εποχή το Ευρωκοινοβούλιο που ανέβαλε τα καθήκοντά του προλίγου και είναι αμέσω κινητοποιημένο, έτοιμο να διαπραγματευτεί, έτοιμο να αναλάβει πλήρω τι ευθύνε του και τα καθήκοντά του. Ξέρουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και είναι συγχρονισμένο με την στατική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η προοπτική μια διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη είναι κάτι που μπορεί να μας επιτρέψει να ανασκουμποθούμε, να αναλάβουμε δράση και να προχωρήσουμε για να πάμε πιο πέρα το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δέκα χρόνια μετά τη συνθήκη της Λης που δεν έχει ακόμα δώσει όλα τα αποτελέσματα που θα μπορούσε. Ας προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο τα δέκα επόμενα χρόνια με αισιοδοξία, ελπίδα και ε, με χαρά χωρίς να ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό όνειρο, το ευρωπαϊκό επίτευγμα πρέπει με ρεαλισμό και πραγματισμό να το φέρουμε εις πέρας, αλλά και με αποφασιστικότητα για να, για να ωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όποια και αν είναι η καταγωγή τους, η υποκότητά τους, η εθνικότητά τους ή οι θρησκευτικέ τους πεπιθήσεις. Αυτές είναι οι βασικές μας αξίες, οι αξίες που ε, δημιουργούν αυτήν την ευρωπαϊκή ψυχή και αυτό το επιπλέον που έχει η ευρωπαϊκή ψυχή. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε με όλους όσοι πήραν το λόγο. Η συζήτηση για το σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ε, θα κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακολουθεί ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου. Θυμίζω ότι μπορείτε να ζητήσετε ε, το λόγο ε, στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ και με τις μπλε κάρτες χρησιμοποιώντας τη συνήθη διαδικασία ή το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά. Δίνω μέσω το λόγο στον πρόεδρο Σάγλ Μισελ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερη τιμή για μένα και προνόμιο ευκαιρία που έχω να παίρνω το λόγο ε, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το νέο θεσμικό κύκλο και θα ήθελα να εκφράσω μια ευκή και ελπίδα να αναπτυχθεί μια ποιοτική θεσμική διοργανική συνεργασία στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την φιλοδοξία. Την φιλοδοξία να συνάψουμε μια ε, συμφωνία ειρήνης με τη φύση. Η κλιματική αλλαγή είναι απειλή. Ε, την έχουμε μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη μεγάλη φιλοδοξία για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Και λίγες ώρες μετά ε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα κατέληξε με στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050. μια χώρα έχει περισσότερο χρόνο ε, να εφαρμόσει ε, αυτά τα θέματα. Είναι ένα τεράστιο άλμα, ομόφωνο, ε, στη σωστή κατεύθυνση για να προχωρήσουμε σε αυτό το εγχείρημα. Είναι σαν να στέλνουμε ξανά έναν άνθρωπο στη σελήνη, έτσι το έχουμε ονομάσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο και αυτή τη δέσμευση και θέλω να τονίσω ότι σωστά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάλαβε ότι αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη από κοινωνική πλευράς και χρειάζεται και επιπλέον πόρους. Εξού και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχει μεγάλη φιλοδοξία για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Ε, πραγματικά χρειάζεται ε, ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης ε, εκτός από το Ταμείο Αλληλεγγύης που πρέπει να καταλάβει ότι δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία όλα τα κράτη-μέλη, ότι οι πραγματικότητες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Για να έχουμε μια στρατηγική που να σέβεται τις επιλογές των διαφόρων κρατών μελών ως προς το ενεργειακό τους μείγμα. Αυτά ως προς το πρώτο σημαντικό θέμα που έχουμε να δώσουμε τη μάχη αυτή κατά της κλιματικής αλλαγής και αυτή τη σοβαρή πρόκληση να την μετατρέψουμε σε πραγματική ευκαιρία έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι ε, ήπειρος ηγέτης σε αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κινητοποιηθεί για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς πολιτικά προς το σκοπό αυτό. Κυρίε και κύριοι, ο επόμενο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι πολύ περίπλοκο. Είναι περίπλοκο θέμα και δύσκολο, γιατί έχουμε ένα χάσμα τώρα, ένα έλλειμμα με το Brexit. Θα πρέπει κάποιε χώρε να πληρώσουν περισσότερα και κάποιε άλλε να ε, λάβουν περισσότερα. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών με σεβασμό για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως απορρέει από τις συνθήκες. Η επόμενη συζήτηση λοιπόν για τον ευρωπαϊκό Προεπολογισμό δεν είναι μόνο ένα θέμα ποσοστού του ΑΕΠ, δεν είναι μόνο ένα θέμα εθνικών συνεισφορών, που προφανώς αυτό βλέπουν τα κράτη-μέλη, αλλά είναι επίσης και ένα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο, με τις προτεραιότητες και με την ουσία. Τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα έτη. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θέλουμε να αναπτύξουμε τα επόμενα έτη. Άλλο σημαντικό θέμα λοιπόν θα είναι η σωστή ισορροπία που θα να βρούμε ανάμεσα στις κλασικές ευρωπαϊκές πολιτικές όπως είναι η γεωργία και η συνοχή από τη μια και από την άλλη τις νέες πολιτικές και τις νέες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, καινοτομία όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με το Κοινοβούλιο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα τους επόμενους μήνες. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ρεσιμότητας. Για διάφορες χώρες αυτό μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Σε κάποια κράτη μιλούμε για κράτος δικαίου, σε κάποια άλλα για τη μετανάστευση, ε, ε, για το κοινωνικό ντάμπινγκ, φορολογικό ντάμπινγκ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για τον προπολογισμό θα είναι η ευελιξία. Υπάρχουν πολλές χώρες, και το κατανοώ, που ζητούν περισσότερη ευελιξία. Θα δούμε τι περιθώριο υπάρχει εκεί για συμβιβασμούς, για όλα αυτά τα θέματα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι φυσικά το ζήτημα των ιδίων πόρων. Σημείωσα πραγματικά στον προπολογισμό κάποια ισχυρά μηνύματα που έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του θέματο. Δηλαδή, όταν γίνεται συζήτηση για αυτά τα σημαντικά θέματα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει μπορεί να διευρυνθεί το σύστημα ETS εμπορίας εκπομπών ρήπων ή θα πρέπει να συνδεθεί με την ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Ή άλλοι προτείνουν φορολογία για τα πλαστικά. Ξέρετε ότι είναι πολλά τα ζητήματα εκεί. Για τη διαδικασία τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Το Συμβούλιο μου έδωσε την εντολή ε, και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσουμε εντατικά τις διμερείς διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη με πρόθεση να ε, προχωρήσουμε προς ένα συμβιβασμό. και να αξιολογήσουμε ποια στιγμή βρισκόμαστε σε μια ζώνη πολιτικής προσγείωσης για να οδηγηθούμε στην τελική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω ε, να έχουμε ε, εκ των προτέρων ε, συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χτες έγινε μια πρώτη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου για να παίξει πλήρως ε, το θεσμικό του ρόλο το Κοινοβούλιο που απορρέει από τη συνθήκη. Πάντα με σεβασμό και με επιθυμία να έχουμε αυτή την αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Σύντομα, ασχοληθήκαμε και με το θέμα του Brexit. Σύντομα. Διότι αυτό το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων ε, της εκλογικής αναμέτρησης και με πολύ μεγάλη νυφαλαιότητα και ηρεμία είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα υπό την αιγίδα του Μισελ Μπαρνιέ